μια ματιά. Είναι ένα βιβλίο τόσο. Γεμάτο τεχνικές ε, λεπτομέρειες ε, και χρειάστηκαν 10 χρόνια για να συμφωνήσουμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολο να φτιάξουμε άλλη μια συμφωνία με τον ίδιο βαθμό περιπλοκότητας σε ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον. Γι' αυτό Πρέπει να επιμείνω ότι για εμάς τους Ευρωπαίους και μιλάω εξ ονόματος του Συμβουλίου Εξωτερικών ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιζήσει αυτή η συμφωνία. Και γι' αυτό πρέπει να επηρεάσουμε τους Ιρανούς για να εκπληρώσουν τις ε, δεσμεύσεις τους. Αλλά να σας πω και κάτι που είχα πει στην αρχή. Οι Αμερικανοί αποσύρθηκαν μόνο μερός από την συμφωνία. Και οι Ιρανοί σέβονταν τις υποχρεώσεις τους ε, επί 14 μήνες χωρίς καμία ε, αντίρρηση. Τώρα βεβαίως είπαν ότι θεωρούν ότι δεν δεσμεύονται πλέον από την συμφωνία αυτή. Αλλά είναι άλλο να μην αισθάνεται κανείς ότι δεσμεύεται και άλλο να αλλάξει ε, πλευρά. Και εκεί πέρα μόνο η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας μπορεί να μας πει εάν και κατά πόσο συνέβη. Και ακριβώς, ε, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, ε, παρακολουθούμε το τι συμβαίνει. Εξάλλου, μέχρι στιγμής είναι έγκυρες οι αναφορές τους. Περισσότερες επαφές λοιπόν και με το Ιράκ και να δούμε όλα τα κομμάτια της πυρηνικής συμφωνίας για να παραμείνει εν ζωή. Μπορώ να μιλήσω και για το αεροπλάνο, το ουκρανικό. Να προσπαθήσω να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα που θέσατε. Αλλά δυστυχώς θα μακρηγορήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας. Είμαι σίγουρος ότι το ζήτημα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Πριν ε, να περάσουμε στο επόμενο σημείο, μια σύντομη ανακοίνωση. Ο κύριος Λάντς Φορμέν ε, θα γίνει μέλο τη ομάδας ECR ε, από την 15η Ιανουαρίου 2020, εγκαταλείποντας τους μη εγγεγραμμένους. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Βίσιλερ Λίμα, ετήσια έκθεση του 2018 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο θέμα αυτό. Να σας ε, υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ζητήσετε το λόγο για το CATSDI και για την πλακάρτα χρησιμοποιώντα το ηλεκτρονικό σύστημα και την πρώτη γραφή. Έχετε στην είσοδο του ημικυκλίου τις οδηγίε. Και τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. κυρία Βίσελη Λίμα, παρακαλώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μιλήσει με ισχυρή, ξεκάθαρη και ενωμένη φωνή όταν μιλάμε για τα ανθρωπίνα δικαιώματα ένα ε, θέμα ε, που ε, πρέπει να καταλήξουμε σε συνένεση και θα εκφράζει όλες τις πεπιθήσεις μας, όλες μας τις μάχες και θα μπορούσε η έκθεση αυτή να εγκριθεί από μεγάλη πλειοψηφία. Ε, το να είμαστε ενωμένοι ε, μας επιτρέπει σε ε, να δηλώσουμε τον βαθύ μας σεβασμό απέναντι στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να υπερβαίνουμε τα σύνορα μεταξύ των κομμάτων όταν πρόκειται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αξιόπιστοι όταν ε, πάντοτε στις διεθνείς μας σχέση ζητάμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αυτή τη φορά όμως ε, είναι ε, κάτι πάνω από υπεράτητο αν δούμε το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης. Η ετήσια έκθεση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία για τις επιθέσεις κατά του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Ένα σημείο που ιδιαίτερα με ανησυχεί είναι η αύξηση του αυτορχισμού ως πολιτικό πρόγραμμα. Ε, επίσης, ε, δεν ε, θέλουμε να πέσουμε στον πεσιμισμό η έκθεση. Εκφράζει την ικανοποίησή τη για το ότι σε ορισμένε χώρε η διαδικασία ειρήνη και εκδικονοτισμού υλοποιείται, καθώ και έχουμε και μεταρρυθμίσει σε συνταγματικό και δικαστικό επίπεδο. Η κοινωνία των πολιτών ε, σήμερα ε, έχει μεγαλύτερη προβολή, ενθαρρυντική προβολή. Εμείς υποστηρίζουμε όσους υπερασπίζουν τις δημοκρατικές αξίες. Όμως ε, έχουμε ένα ιδιαίτερα ζωφερό σημείο για την ανθρωπότητα η μάστιγα των σειράξεων ε, και της εθνοκάθαρσης συνεχίζει ε, να οδηγεί στο θάνατο πολλούς ανθρώπους ε, και να προκαλεί μαζικούς εκτοπισμούς και συχνά έχουμε απάνθρωπες δράσεις από την πλευρά των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν αυτός ο χώρος γίνεται ένας χώρος καθημερινής σκληρότητας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 ο καθένας από μας, όλοι μας, υποχρεούμαστε ως άνθρωποι να το καταγγέλουμε αυτό με την φωνή και ως μέλη του Κοινοβουλίου έχουμε την πολιτική υποχρέωση να προκαλέσουμε τη δράση κατά της ανθρώπινης εξαθλίωσης. Η έκθεση αναφέρεται επίσης ε, στα δικαιώματα των ε, αυτόχθονων πληθυσμών. Υπογραμμίζει το ότι πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα των φίλων. Οι γυναίκες και τα παιδιά βρίσκονται ε, σε ευαίσθητα περιβάλλοντα και ε, πολύ συχνά είναι οι πληθυσμοί που υφίσταται τις ε, περισσότερες οδικίες. Ε, επίσης, ε, αναφέρεται η έκθεση και στο πληρισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρεται στις οδικίες κατά των υπερσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταδικάζει την θανατική ποινή, τις διώξεις, τις αυθαίρετες και ε, επίσης δηλώνει ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ενισχύονται. Υποστηρίζει πλήρω το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τι τρίτε χώρε ε, για την πρόθεση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, υπογραμμίζει ότι η ελευθερία τη συνείδηση, ε, τη θρησκευτική πίστη και πεποίθηση θα πρέπει να είναι αντικείμενο εγγύηση σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω το σύνολο των σκιώδων εισηγητών ε, και των ομάδων τους ε, για το επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα το εκπρόσωπο, κύριο Μπορέλ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με και πάλι θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ανά τον κόσμο. Χαιρετίζω την εμπεριστατωμένη αυτή ετήσια έκθεση ε, που παρέχει πολλές χρήσιμες συστάσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, κυρία Ιζαμπέλο Άιζερ Βάισλερ Λίμα για το έργο της. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των προσπαθειών μας γιατί αποτελούν τμήμα του DNA μας. Στην ε, πρώτη συμφωνία, συγγνώμη, στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών, ε, το οποίο προείδρευσα το Δεκέμβριο, συζητήσαμε τι συλλογικέ μα προσπάθειε για να προαγάγουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα για τη δημοκρατία, λαμβάνοντα υπόψη τι ανησυχητικέ ε, τάσει που παρατηρούνται με τις αυξανόμενες επιθέσεις προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το καθεξής. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το καθεστώς κυρώσεων για την κατάλυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει όλοι μαζί και θέλουμε να τον επιτύχουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Τη δεύτερη μέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ήρθα σε επαφή με οι υπερασπιστές ε, των ανθρωπινών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στο Φόρουμ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκεί συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Πολλά από τα ζητήματα που θίξατε στην ετήσια έκθεσή σας, η οποία υιοθετήθηκε το Μάιο, ε, είχαν ήδη ε, εξεταστεί. Εμείς ε, στην δική μας έκθεση χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα παραδείγματα αναχώρα. Ε, έχουμε πλήρη επίγνωση της ισχυρής διασύνδεσης μεταξύ των δύο εκθέσεων. Και για την επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 θέλουμε να υπάρξει έγκαιρα έγκρισή της ε, την Άνοιξη. Στην έκθεσή σας ζητάτε ε, μία βελτιωμένη ε, πολιτική ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό εντάσσεται στο νέο σχέδιο δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Θα είναι ένα οδικό χάρτη που θα θέτει τι φιλοδοξίε και προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πεδίο για τα επόμενα πέντε έτη και θα προβλέπει μία μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο και την αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι και θα πρέπει να παραμείνουν λοιπόν στο επίκεντρο των σχέσεών μας με τρίτες χώρες. Ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι το μεγαλύτερο δημοσιονομικό, ε, μεγαλύτερο δημοσιονομικός μηχανισμός στον κόσμο ε, που αφορά συγκεκριμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. 135 εκατομμύρια διατέθηκαν το 2018 υπό αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Το 2018 είχαμε μία πρόσκληση υποβολής ε, προτάσεων που οδήγησε στην επιλογή πέντε έργων για τα δικαιώματα των ατόμων ε, ΛΟΑΤΚΙ με χρηματοδότηση 70 εκατομμύρια. Ε, αυτό κάλυψε συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν δυσκολίες, Ρωσία, ε, Μαλάου, Νικαράγουα, Ανδόρα, Περού και άλλες. Και εκεί στηρίξαμε την οικοδόμηση δυνατοτήτων και παρήχαμε νομική συνδρομή στα θύματα ε, επιθέσεων κατά τον ΛΟΑΤΚΙ και υπερασπιστήκαμε όσους υπεραμείνονται αυτών των δικαιωμάτων. Η έκθεσή σας πολύ σωστά παρατηρεί ότι το εμπόριο και οι οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να συνδέονται με το πολιτικό διάλογο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε οποιαδήποτε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζετε πολύ καλά τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ε, υπάρχει διάλογος και διπλωματία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε και τον ε, αρμόδιο εκπρόσωπό μας και υπό τη δική του ηγεσία έχουμε αυξήσει σημαντικά την προβολή των θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτική μας. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στην ε, προαγωγή των ε, ε, δικαιωμάτων του παιδιού και μαζί και με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής έχουμε υποβάλει προτάσεις. Δύο παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ένα αφορούσε τα δικαιώματα του παιδιού και το δεύτερο αφορούσε τα παιδιά με αναπηρίες ε, και σε σχέση με το δικαίωμα στην ε, εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και αποκλήσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Σωστά επίσης παρατηρήσατε ότι υπάρχει επαναχώρηση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διατηρεί την προσήλωσή της ε, στην ε, πλήρη περάσπιση των δικαιωμάτων από όλους. Ιδίω ό,τι αφορά τι γυναίκε ε, είχαμε και την πρωτοβουλία για να τεθεί ένα τέλος ε, στο φαινόμενο της βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών ε, τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Αυτή η πρωτοβουλία τη χάνει τη στήριξη σε μιας επένδυσης 500 εκατομμυρίων σε μια περίοδο από το 2018 μέχρι το 2024. Δύο πυλώνες έχουν υλοποιηθεί παραμένει ένας, ε, μάλλον ο ένας πυλώνας αφορούσε ε, ε, τα εγκλήματα κατά των γυναικών και ο άλλος την σεξουαλική παρενόχληση. Όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών μας, ιδίως και εν ώψη της 25ης επαιτίου της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις γυναίκες και την διακήρυξη του Πεκίνου. Η έκθεσή σα χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Δημοκρατία τον περασμένο Οκτώβριο και επισημαίνει την σημασία των διαφανών, συμπεριληπτικών και αξιόπιστων εκλογών. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη, καθώς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ε, συμμετείχαν στις ε, αποστολές εκλογικών παρατηρητών. Πρόκειται για ένα θετικό παράδειγμα που δείχνει ε, πώς μπορεί να υπάρξει σωστή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δεν θέλω τώρα να διατρέξω τον κατάλογο αυτών των αποστολών. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο κάποια. Σαλβαδόρ, Κοσφοπέδιο, Μαλάουι, Σρι την Ισία και άλλες τέτοιε αποστολέ είχαμε. Λυπάμαι που δεν ήμασταν στι τελευταίε εκλογές στη Βολιβία. Θα το διορθώσουμε αυτό και θα συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για να υπερασπιστούμε τη βάση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι μια αποτελεσματική δημοκρατία. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων ήταν πολύ χρήσιμη. Και κλείνοντας θα πω ότι είμαι βέβαιος πως ακούγοντάς σας, ε, κυρία εισηγήτρια, ακούω στα λόγια σας και στο έργο σας ε, τον ίδιο σκοπό που έχει και η υπηρεσία μας. Και έχουμε από κοινού την ευθύνη να εργαστούμε σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έχετε κάνει. Τώρα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι ζητάτε από την Υπηρεσία εξωτερική δράση σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, γιατί εσείς ως Ευρωβουλευτές και εμείς, καθώς εργαζόμαστε στις αποστολές μας σε όλο τον κόσμο, παλεύουμε για τους ίδιους σκοπούς. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Τόματς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Μπορέλ, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πρόκειται για μια πολύ καλή έκθεση που δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε για να υπερασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο θα περιοριστώ σε ένα θεμελιώδες ε, ε, δικαίωμα που μας κάνει να έχουμε μεγάλη επιρροή, να έχουμε μεγάλη επιρροή στον κόσμο, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Κύριε Μπορέλ, ζητώ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να κάνει περισσότερα για να υπερασπίσει χρησιμοποιήσει την ελευθερία της έκφρασης ε, στις γειτονικέ μας ε, χώρες. Ε, είναι πραγματικά παράδεκτο στην Τουρκία να κλείνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, να απολύονται χιλιάδες δημοσιογράφοι και κάποιοι να συλλαμβάνονται και να φυλακίζονται δίκως. Πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση να παραμείνει πραγματικά θεμελιώδες δικαίωμα στη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κύριο Κοτσολίνο, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν ε, είναι κάτι τελετουργικό, ε, ούτε ε, κάτι γραφειοκρατικό αυτό που συζητάμε σήμερα. Η ψηφοφορία όμως και η έγκριση έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση, με 1,5 χρόνο καθυστέρηση. Η δουλειά που κάναμε μας επέτρεψε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε πάρα πολλά θέματα και θα ξέρουν ποιε είναι οι κοινοτομίε τη έκθεση οι συνάδελφοι. όμω εγώ θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι δώσαμε πολύ έμφαση για το πώ θα κάνουμε πιο αποτελεσματική την ευρωπαϊκή πολιτική για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Είναι ένα ουσιώδε θέμα. Ε, που προσπαθήσαμε να θέσουμε στο επίκεντρο απέναντι ε, στην πρόκληση της ε, υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Αυτή είναι η δουλειά και η ευθύνη μας και θα πρέπει στις επόμενες εκθέσεις να μπούμε στην ουσία. Ε, αυτό ε, πρέπει να το καταστήσουμε πραγματικά κεντρικό ζήτημα χωρίς μεν και αλλά. Και θα πρέπει να κάνουμε και κάσσερες προσπάθειες στην επόμενη G20 έτσι ώστε να βάλουμε κάποιους όρους στη συμμετοχή μας και να θέσουμε το μεγάλο ζήτημα των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του Renew, ο κύριος Γκερέντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ετήσια συζήτηση που έχουμε για την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει ένα κίνδυνο να γίνουν οι συζητήσεις μας συζητήσεις ε, ρουτίνας όταν μιλάμε για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, παγκοσμίω. Ε, και ε, μπορεί να προσφεύγουμε σε παρόμοιες ε, διατυπώσεις και να ανανεώνουμε τις ίδιες ελπίδες. Όμως ε, σήμερα είναι διαφορετική κατάσταση. Έχουμε μια καλή έκθεση ενώπιών μας με πολύ καλή δομή και είναι πάρα πολύ ακριβή. η έκθεση που μας παρουσίασε η κυρία Βίσλερ Λίμα είναι ε, πραγματικά σημείο αναφοράς ε, για ε, τους επόμενους μήνες και ίσως και έτη. Πραγματικά προσεγγίζει όλα τα θέματα χωρίς να χάνεται υπερβολικά στις λεπτομέρειες. Επίσης, θήτης βαριές τάσεις που αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Ε, βέβαια μεταξύ αυτών των τάσεων ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και η παναχώρηση της ε, πολυμέρειας. Εγκαταλείπουμε ένα κεκτημένο ότι αφορά το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όποιος παραχωρεί από την πολυμέρεια διαπιστώνουμε παράλληλα ότι κάποια κράτη του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν παρασυρθεί προς αυτήν ε, την κατεύθυνση. Και λυπάμαι πολύ που μεταξύ αυτών έχουμε και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μας πει ποια συνέχεια επιφυλάσσει στις προτάσεις μας. Πέρσι παρουσίασα μία έκθεση για την απαγόρευση των καταναγκαστικών ε, γάμων και των γάμων ανηλίκων. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία ε, την ε, απαγόρευση των γάμων ανηλίκων, των καταναγκαστικών γάμων ανηλίκων και αποφασίσαμε αυτό να το εντάξουμε ως προϋπόθεση στις εξωτερική μας σχέση. Η τελευταία λέξη όμως δεν έχει ακόμα υποθεί. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα την κυρία Νόιμαν για τους πράσινους ένα λεπτό. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χειροτερεύει παγκοσμίω. Γι' αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχει στην διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση με την οικονομική μας δύναμη για να προστατεύσουμε αυτούς που παλεύουν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί μπορούμε να προστατεύσουμε επιχειρήσεις αλλά όχι ανθρώπους. Γιατί εξακολουθούν να πλουτίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πουλτίζοντας όπλα. Πουλώντας όπλα, με Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν χρειάζονται προστασία και γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείε καταστρέφουν το βιός τόσων ε, αυτοχθώνων ανθρώπων για να εξορίξουν άνθρακα. Κύριε Μπορέλ, θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα με αυτήν την έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο και ελπίζω να σας καθοδηγεί στα επόμενα πέντε χρόνια. Και σας ευχαριστώ, κυρία Βίζελερ Ντελίμα, για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπαλντασάρε για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα είμαι εδώ πέρα για να σας ε, παρακαλέσω να μην είστε συνένοχοι σε μια εσχρή υπόθεση εκατομμυρίων δολαρίων, την παρένθετη μητρότητα. Πλούσιοι δυτικοί εκμεταλλεύονται γυναίκες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Πρόκειται για μια νέα μορφή απεικιοκρατίας ή ακόμα χειρότερα σκλαβιάς παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια της γυναίκας και του σώματός της. Ε, παιδιά που τα παίρνουν από τις ε, μητέρες της ή γίνονται αντικείμενο σύμβασης, παραβιάζοντας και την ε, σύμβαση για την, τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και τις σχετικές συμβάσεις για την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος. Η προστασία της γυναίκας λοιπόν δεν πρέπει να παραμείνει να κούφια λόγια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε ό,τι μπορείτε για να σταματήσει η παρένθετη μητρότητα. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για γυναίκες. Οι γυναίκες δεν είναι θερμοκοιτίδες, ούτε τα παιδιά είναι εμπόρευμα. Σας ευχαριστώ. Τσαρνέτσκι τώρα για ένα λεπτό για την ομάδα. ECR. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε. Τα δύο τρίτα της ομιλίας σας, ε, οι οθόνες έδειχναν ε, ότι μιλάτε στην συζήτηση για το Ιράν και το Ιράκ, αλλά κατά λάθο έγινε αυτό. Έλαβα όμω μήνυμα που έλεγε ότι είναι περίεργο, γι' αυτό το αναφέρω. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε το θεσμικό όργανο που ε, δίνει το σωστό δημοκρατικό παράδειγμα στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Και αυτό είναι θετικό. Έχω υπάρξει παρατηρητή ε, κατά τη διάρκεια εκλογών σε 20 διαφορετικές χώρες και ξέρω ότι ε, είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι αποστολές. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, έχει έτσι κατάσταση, ώστε εμείς να πρέπει να διατηρούμε κάποια δημοκρατικά πρότυπα. Και το λέω γιατί έχω λάβει πληροφορίες. Δώστε μου λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί μιλούσα για την οθόνη προηγουμένως. Λοιπόν, χθες ε, δεν υπήρξε τελικά συζήτηση για τα όσα συνέβησαν στο Παρίσι. Και διακόπτεται το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο για ένα λεπτό. Για την ε, Γκουέντζιελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2018 Είδαμε μίσος, μισαλοδοξία, αυξήθηκε η πολιτική βίω κατά των υπερασπιστών, των δικαιωμάτων ε, και του περιβάλλοντος. Ε, Παραδείγματο χάρη η Μαριέλ Φράγκο δολοφονηθήκε. Εξακολουθούμε να ζητάμε δικαιοσύνη σήμερα. Όμως επίσης ήταν το έτος που οι γυναίκες βγήκαν μαζικά στους δρόμους να μας υπενθυμίσουν ότι η Επανάσταση θα είναι φεμινιστική, δεν θα γίνει καθόλου. Και ένα έτος μετά η έκθεση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα αρνείται ε, να εξετάσει την Ευρώπη και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και εδώ παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ας δούμε τι συμβαίνει στα σύνορά μας, ε, στη Μόρια. Ε, έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκά Γουαντάναμο όπου η ανισότητα βασιλεύει. Ακόμη και στους δρόμους μας απαιτούμε υποκριτικά πολλές χώρες να γιώνται τη σοβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενώ εμείς επιτρέπουμε στις πολυεθνικές μας να τα παραβιάζουν. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Πρέπει να σταματήσουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Ευρώπη και επίσης από ε, τις κυβερνήσεις και τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική. Ευχαριστώ. Καστάλντο για τους μη εγγεγραμμένους για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα ψηφίσουμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Πρόκειται για κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη μία φορά πρέπει να επιβεβαιώσουμε την σημασία των θεμελιωδών αυτών αξιών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολυμέρεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα θυμίζει το τι μπορούμε να κάνουμε εάν ε, οι δράσεις μας βασίζονται σε αυτές τις αρχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Βίζελερ Λίμα, για το ότι συγκέντρωσε τα, τις διάφορες απόψεις στην έκθεσή της. Το στρατηγικό αυτό έγγραφο παρουσιάζει την βαθύτατη ανησυχία που έχουμε όλοι μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Το 2019 ήταν ένα έτος όπου είδαμε όλο και μεγαλύτερες ε, και ανησυχητικότερες τάσεις ε, προς την αυταρχικότητα. Αυτή τη στιγμή πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να ζητήσουμε και όλοι οι υπόλοιποι να σέβονται τους κοινούς κανόνες. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στον κύριο Φαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περιμένω γιατί ασχολείται με το τηλέφωνό του ο κύριος ε, Μπορέλα. Τουλάχιστον να βάλει τα ακουστικά του. Δυστυχώς ε, είναι αναγκαίο στην έκθεση αυτή την οποία έχουμε μπροστά μας να αναφερθούμε σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον κόσμο δισεκατομμύρια άνθρωποι θέλουν να μπορούν να μιλούν ελεύθεροι. Δυστυχώς όμως ε, αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες, ε, φυλακίσεις μέχρι και δολοφονούνται. Έχουμε λοιπόν ε, καταπίεση, καταστολή δολοφονίες στο Ιράν, στην Ινδία, Νεπάλ, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Σομαλία και ελπίζω να αφήσει κάποτε κάτω το τηλεφωνό του ο κύριος Μπορέλ. Η ευρωπαϊκή πολιτική λοιπόν είναι δυτή. Αφενός καταδικάζουμε αυτά και δικαίως. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει πολύ επικερδές εμπόριο με αυτές τις ε, χώρες. Οπότε εδώ πέρα απαιτούνται συγκεκριμένες πράξεις γιατί τα ωραία λόγια χωρίς πράξεις είναι κούφια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον... την κυρία Σάντος. Η παρουσίαση της έκθεσης αυτής ε, δεν είναι απλή υποχρέωση, ούτε είναι γραφειοκρατική τελετουργία. Έχει προκύψει από βαθύ προβληματισμό και σκληρή δουλειά, διαλόγου και συντονισμού και ε, απαιτεί συγκεκριμένη εφαρμογή στην καθημερινή ζωή ανθρώπων. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια αλλά και το σκιώδη εισηγητή της ομάδας μας, τον Αντρέα Κοτσολίνο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 επειδή δεν έχω χρόνο, θα αναφερθώ απλώ σε κάποια σημεία τη ε, έκθεση. η ε, σημασία που δίνεται στην, στο ρόλο τη ε, κοινωνία των πολιτών, το ότι υπογραμμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί η ελευθερία τη έκφραση και τη δημοκρατία σε περίοδο μεγάλων προκλήσεων. Η αναφορά στο να ενισχυθεί η καταπολέμηση τη ατιμορρησία, η αναγκαιότητα τη προστασία των αυτόχθων λαών που εκτίθενται, λένε και περισσότερο, σε κάθε πηγή. Επίση ε, Επίσης, ε, να αναφερόμαστε στου εκτοπισμένου. Ε, Ξεπέρασαμε τα 80 εκατομμύρια πέρσι. Η αναφορά που γίνεται στην ισότητα των φύλων και στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε πολύ περισσότερα που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Ας είναι αυτή η κινητήρια δύναμη τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Φον Βίζε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ξέρετε πού κατασκευάστηκαν οι κάρτε που στείλατε τα Χριστούγεννα. Το Δεκέμβριο, ένα κορίτσι στον βασίλιο Βασίλειο βρήκε ένα μήνυμα σε μια ευχετήρια κάρτα, ε, ένα μήνυμα που ζητούσε βοήθεια. Ήταν από το άτομο που αναγκάστηκε και καταναγκάστηκε να ε, φτιάξει αυτή την κάρτα σε ένα κελί φυλακών στην Κίνα. Οι πλουσιότερες ε, χώρες του κόσμου έχουν ε, πρόσβαση σε πολύ φτηνά τέτοια προϊόντα και γυρίζουν ε, την πλάτη στο πραγματικό ανθρώπινο κόστος. η πολιτική είναι δεν γνωρίζουμε και ούτε θέλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει ε, στην, ε, στο κάτω μέρος της γραμμής ε, ανεφοδιασμού. Αυτή είναι η πολιτική των πολυεθνικών του λιανικού εμπορίου. Πρέπει η ιδέωσα επιμέλεια να γίνει υποχρεωτική. Οι εταιρείε να διασφαλίζουν ότι η χαμηλή τιμή των προϊόντων τους δεν έρχεται και δεν εξασφαλίζεται σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Χάουταλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Πατεκπρόσωπε, ήθελα να επισημάνω ε, το ισχυρό μήνυμα για την ισχυρή έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να θεσπιστεί ιδέως επιμέλεια για τις επιχειρήσεις σε ό,τι φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εταιρείε ε, πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Και χαίρομαι που όλα ένα και περισσότερες εταιρείε ζητούν τη θέσπιση αυτών των διατάξεων, ιδίω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί θέλουν ίσο πεδίο ανταγωνισμού. Να μην ε, τους διώξουν από την αγορά άλλε άλλε ανεύθυνες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν ε, να ενθαρρύνουμε την υπευθυνότητα και όχι την ανευθυνότητα. Είναι σημαντικό επίσης να ε, διασφαλίσουμε την πρόσβαση ε, στην, σε ένδικα μέσα προς θύματα τέτοιων πρακτικών και αυτό είναι ο τρίτος πυλώνας του Οδηγού των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ελάχιστα σε αυτό το πλαίσιο. Το 2020 θα πρέπει να είναι η χρονιά που θα αναλάβουμε δράση ε, και να έχουμε ενέργειες που θα έχουν επίπτωση σε πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Ράσεν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές χώρες ακόμα καταπατώνται συστηματικά. Οι προσπάθειε λοιπόν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελούν αιχμή τη εξωτερική μα πολιτική. Και εδώ εννοώ την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των ατόμων με αναπηρία. Σκέφτομαι την δίωξη και βία κατά ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, είτε εξαιτία τη ε, θρησκείας του, της εθνικότητάς του ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Εν τω μεταξύ, θέλω να επισημάνω ότι οι χριστιανοί είναι αυτοί που διώκονται περισσότερο στη θρησκευτική ομάδα από οποιαδήποτε άλλη. Ε, τι έχει να πει ο εξειδικευμένο θεσμικό φορέα Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θρησκευτική ελευθερία. Θα πρέπει να ε, ενισχυθεί και να αυξήσει τι προσπαθίε του και θα ήθελα ο ύποπτο εκπρόσωπο να μα ενημερώσει για την εντολή αυτού του θεσμικού εργάνου για την ε, θρησκευτική ελευθερία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κομίν ή Ολιβέρες για ένα λεπτό. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Εισηγήτρια. Όλοι συμφωνούμε ότι η σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνέ επίπεδο θα πρέπει να βασίζεται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά πώς η Ένωση μπορεί να έχει ε, την ε, ηθική εξουσία ε, για να απαιτεί από τα άλλα κράτη να σέβονται τα δικαιώματα, να έχουμε κράτη-μέλη που δεν είναι ικανά να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο δικό, στη δική τους επικράτεια. Μιλάμε για τα πολιτικά ε, δικαιώματα, τα οικονομικά, εργασιακά δικαιώματα. Ε, δεν ε, έχουν συγκίνηση σεβαστά τα πολιτικά δικαιώματα, γιατί εγώ, παραδείγματο χάρη ο ίδιος, είμαι εξόριστος σήμερα στο Βέλγιο, γιατί δεν σέβεται τα δικαιώματα των Καταλωνών αυτανομιστών. Ε, όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφει το βλέμμα της αλλού, όταν ένα κράτος μέλος ε, παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε ε, χάνει κάθε ικανότητα για να ζητήσει από τους άλλους να σέβονται αυτά που δεν σέβονται τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Um, Υπάρχει μία ερώτηση, μία μπλε κάρτα. Την δέχεστε, 30 δευτερόλεπτα. No, he doesn't accept. I'm sorry. Δεν το δέχεστε, μάλιστα. Με την κυρία Αρενά, για ένα λεπτό. Πίστευα ότι δεν είναι η σειρά μου, γιατί λέει κοκαλάρι στον πίνακα. Α, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Ναι, η κυρία Κοκαλάρη έχει το λόγο. Για ένα λεπτό επίσης. Συγγνώμη, σας παρέλειψα όταν υπήρξε το αίτημα για την πλεκάρτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι η δημοκρατία στον κόσμο υπαναχωρεί και υπάρχει καταστολή των ελεύθερων μέσων περισκής ενημέρωσης. Ε, η βία κατά των ε, γυναικών ε, είναι το πιο κοινό φαινόμενο βίας. Επίσης, βλέπουμε τι συμβαίνει στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Θα ήθελα η Κομισιόν να ασχοληθεί με τρία σημαντικά πράγματα. Καταρχήν, θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις κατά ανθρώπων ε, που προβαίνουν ε, σε μεγάλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και κατόπιν ε, θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρά κριτηρία για τις ε, χώρες προσχώρησης. Θα πρέπει να δώσουμε όμως ε, στις χώρες αυτές ελπίδα το μέλλον τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι αλλού. Και επίση θα πρέπει να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών παγκοσμίω. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ιδέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Αυτό είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στάση και να πούμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό για μας. Μάλιστα, τώρα κύριε Ρενά, για ένα λεπτό. 70 χρόνια μετά από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ζούμε σε έναν κόσμο που ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σε κίνδυνο. Είναι πραγματικά ανησυχητή η έκθεση, σειράξει ε, παντού στον κόσμο στερούν εκατομμύρια ανθρώπους από τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ε, ε, και η άγρια παγκοσμιοποίηση θυσιάζει εκατομμύρια ανθρώπους στο ε, βωμό των μετόχων χωρίς να μιλήσουμε για αυτά αρχικά καθεστώτες που ασκούν καταστολή, διακρίσεις στο όνομα μιας φερόμενης εθνικής ταυτότητας. Όμως και η Ευρώπη βιώνει τέτοια φαινόμενα. Όμως βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά για πόσο καιρό ακόμα είναι το δικαίωμα σε ευθύνη και αφορά και την αξιοπιστία μα ε, να προωθούμε παγκοσμίω τα ανθρώπινα δικαιώματα με συνεκτικό τρόπο όμω σε όλε μα τι πολιτικέ. εμπορική, διπλωματική, πολιτική, στι συμφωνίες σύνδεση. θα πρέπει να θέσουμε σε προτεραιότητα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ε, μείνουν ε, ευρωπαϊκό πολιτικό μήνυμα και εμεί θα σα υποστηρίξουμε κύριε μπορέλε σε αυτό το ευγενέ καθήκον που έχετε αναλάβει σήμερα. Σα ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Ροντρίγκε Ράμο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κουμίν, στις δημοκρατίες όπως στη χώρα μου στην Ισπανία τα ανθρώπινα δικαιώματα αξίζουν αυτό που αξίζουν και ισχύουν. Ε, και ο σεβασμός ε, των αποφάσεων ε, των δικαστηρίων είναι η καλύτερη εγγύηση. Όταν ο σύντροφός σας στράφηκε κατά του κράτους δικαίου στην Ισπανία, παραβίασε τα δικαιώματα των κατολωνών πολιτών, γιατί ως πρόεδρος της κοινότητας αυτής είχε υποχρέωση να τα σέβεται και να τα προστατεύει. Ε, σήμερα διαφεύγει από την Ισπανική δικαιοσύνη για να μην απαντήσει για την πράξη του και κάθεται σε αυτή την έντρα ε, και ε, ουσιαστικά παραγνωρίζει το κράτος δικαίου και αναζητεί ατιμορρησία και όχι ασυλία. Αυτή είναι η περάσπιση των δημοκρατιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Μπρικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, για την εξαιρετική αυτή έκθεση που ελπίζω να υπερψηφιστεί με μεγάλη διαφορά στην Ολομέλεια που μιλά για την ελευθερία έκφρασης, ε, την πολυμέρεια στα μέσα ενημέρωσης και δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή την διατήρηση της τάξης. Έχουμε να κάνουμε και με τις παράνομες κρατήσεις ε, και το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, προαγάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο μέσω της εξωτερικής ε, πολιτικής μας και να μην αφήνουμε κατά μέρο τα πολυτερχικά καθεστώτα. Βέβαια όλα αυτά θα ε, δοκιμαστούν τον επόμενο μήνα, γιατί εκεί θα πρέπει να εκυρώσουμε την εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική παναχώρηση ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ενισχύθηκε αυτή η προβληματική ε, το 2019 πρέπει να αντιδράσουμε σε ό,τι αφορά την κράτηση, τη σύλληψη και κράτηση δημοσιογράφων και blogger. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπεί σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο πλαίσιο τη εμπορική μα πολιτική. Ευχαριστώ, Fitzgerald, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Βίσλερ Λίμα, για αυτή την έκθεση. Όπω έχουν πει και οι άλλοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένη ε, και αποτελεί, πραγματικό παράδειγμα σε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα το ζήτημα είναι πώ θα υλοποιηθεί έχει θέση και έχει αποσταλεί μάλλον σε μια σειρά ε, σημαντικά θεσμικά όργανα και άτομα. Ε, ας κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να υλοποιηθεί στην πράξη προ όφελο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία τώρα κινδυνεύονται. Και έχουμε και αυτή την ε, ε, μάτσο ηγεσία σε διάφορες χώρες του κόσμου. Πρέπει εμεί λοιπόν να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών μετά και από την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και έχουμε μάλιστα και έξι χώρες που δεν την έχουν κυρώσει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταργηθεί ο ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να υπερασπιστούμε του ε, υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. έστερα για ένα λεπτό. Στο άρθρο 2 της Σύμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, κράτος δικαίου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν δεν ισχύουν μόνο για τους πολίτες της Ένωσης αλλά ανεξαιρέτως για όλους αλλά σε τι χρησιμεύουν σε έναν πρόσφυγα που έχει κολλήσει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και για νιωστή φορά τον αποθούν οι κροατικές αρχές παρανόμως και τον, εκεί πέρα τον δέρνουν και τον κλέβουν. Κυριολεκτικά τους πατάνε με τα πόδια και από ό,τι φαίνεται το, αυτό το οποίο παίζει τον κύριο ρόλο στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης είναι η απόκρουση των προσφύγων. Και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το δικαίωμα στο άσυλο και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Σάντσε Σαμόρ. Ευχαριστώ. Καθώς ο κύριος Κουμίν ε, δεν είχε το θέλος να δεχτεί την μπλε κάρτα, Θέλω, θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό το έγγραφο αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Περιμένω χάρη στι 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017, αυτό που έκανε το Καταλληνικό Δικοινοβούλιο, όταν καταπατήθηκαν τα δικαιώματα τη μειονότητα. Το ίδιο δικαίωμα ε, που έχει ο κύριος Κουμέιν, ε, που κάθεται εδώ, όλοι όσοι είμαστε εδώ ε, σεβόμαστε όταν μας αποδίδουν το δίκαιο ή όχι. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο ξέρετο έργο της εισηγήτριας ε, ε, και ε, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν είναι παγκόσμιος παίκτη μόνο απονέμοντα το βραβείο Σαχάροφ. Εμεί έχουμε την ικανότητα και την επιρροή παγκοσμίω. Θα πρέπει η δική μας πολιτική πρόθεση των αξιών να συνοδεύεται από και μια πολιτική υπεράσπισης των αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων στα καθεστώτα που δέχονται επίθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόλατ για ένα λεπτό. Σας είδα. Τώρα πριν από λίγο την είδα. Δεν είναι εδώ. Συνεχίζω με το KCI. Συγγνώμη, πέντε συναδέλφους θα δεχτώ μόνο. Προσπαθώ να σέβομαι όλες τις ομάδες. Ξεκινάμε τον κύριο Πόσφυσιλ. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε εκπρόσωπε, έχω ένα σχόλιο για τη συζήτηση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά είναι αντικείμενο συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συχνά συζητάμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες περιοχές ε, στον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να καλέσω η έκθεση αυτή να αποτελέσει κατευθυντήρια γραμμή ε, στην εξωτερική μας πολιτική. Συνεχώς ε, μιλάμε για την αποφυγή της ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να είμαστε πιο αυστηροί απέναντι σε χώρε και περιοχέ που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήθελα εμείς ε, να υλοποιήσουμε την υπόσχεση αυτή, θα ήθελα εμείς να αναλάβουμε δράση κατά τον ίδιο τρόπο και θα ήθελα εμείς να υποστηρίξουμε τα κράτη που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεχίζουμε με την κυρία Βάρτ ε, για ένα λεπτό. Η έκθεση αυτή επαναλαμβάνει και στηρίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περάσαμε τον Μάιο του 2018 όσον αφορά την προστασία των παιδιών μεταναστών. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε τις ε, σχετικές προτάσεις στην ε, Συμφωνία για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για προδοσία της ε, δέσμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου για ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήθελα να επενέσω τον Λόρδο Ντάμπς, ο ίδιος ε, γιος ε, Εβραίων ε, προσφύγων που επέκρινε την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης. Αν αυτή είναι η παγκόσμια Βρετανία στέλνει λάθος μηνύματα για το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να είμαστε. Είτε εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις δεσμεύσει μας ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εγώ ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων του παιδιού θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους κρατούντες να θυμηθούν τον Άλαν Κέρντι και τα άλλα παιδιά πρόσφυγες που πέθαναν. Σας ευχαριστώ. Αουστρεβίτσιους για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Παρά τις ε, προσπάθειες, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν βελτιώνεται τα εγκλήματα κατά γυναικών, παιδιών, μειονοτήτων, θρησκευτικών ομάδων. Ε, είναι δύσκολο να τα αντιληφθούμε, ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε επί σειρά ετών με αυτά τα ζητήματα. Το ερώτημα του εάν η αξιολόγηση και η αντίδρασή μας είναι η καλύτερη παραμένει ανοιχτό. Παραδείγματο χάρη, ανεδρούμε πάρα πολύ αργά στην κατάσταση στην Καμπότζη, όπου οι επιθέσεις ε, στην αντιπολίτευση, στην κοινωνία των πολιτών και στα μήμια έχουν ενταθεί. Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης λαμβάνουν χώρα και κοντά στα σύνορά μας. Στη Λευκορωσία δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση στις ε, πολιτικές διαδικασίες μεταξύ των οποίων η ελευθερία του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε, η ελευθερία λόγου και τα ανεξάρτητα μημία. Η πολιτική αντιπολίτευση καταστέλλεται και η κοινωνία των πολιτών παραμερίζεται από τις ε, διαπραγματεύσεις για το να απομακρυνθεί η χώρα από την Ρωσία. Σας ευχαριστώ. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έχουμε τον κύριο Γόλας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιοι λένε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται υπό απειλή. Ισχύει αυτό όμω. Ε, Δυστυχώ έχουμε χάσει το ηθικό πλεονέκτημα να μπορούμε να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω μπορούσαμε παλιότερα. Μόνο και μόνο το γεγονό ότι αγνοούμε το κράτο δικαίου τόσο συχνά σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα ε, δεν αυξάνει την οξιοπιστία μας για να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Το γεγονός και μόνο ότι δεν ε, αντιτιθέμεθα στις αμερικανικές κυρώσεις ε, στο Ιράν, στη Συρία και στη Βενεζουέλα, γιατί οι κυρώσεις αυτές τρέφονται κατά των φτωχότερων και η Ευρώπη θα πρέπει να αντισταθεί. Μιλούμε για εμπόριο και ανθρώπινα δικαιώματα και ότι το ένα ενισχύει το άλλο. Στη Σαουδική Αραβία όμως ε, έχουμε συστηματικά αποκεφαλισμούς ανθρώπων, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εταιρικέ σχέσεις ούτε με το Ισραήλ, παρά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου ε, απέναντι στην Παλαιστίνη συστηματικά. Δεν είμαστε λοιπόν συνεπείς ε, στη συμπεριφορά μας. Ευχαριστώ και επανερχόμαστε στην Κομισιόν. Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπο, έχετε το λόγο. Human rights endless... Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ατελείωτο θέμα. Υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τον ειδικό απεσταλμένο μας για την ε, ελευθερία πεπιθήσεων. Πράγματι έχουμε ένα τέτοιο ειδικό απεσταλμένο, το Ζαν Φίγκελ. Είναι μια θέση που δημιουργήθηκε υπό τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ το 2016 Υποστηρίζει λοιπόν την υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και προστασία των, της ελευθερίας επεπιθύσεων. Αυτό αναφέρεται στην εντολή του. Επισκέπτεται χώρες όπου η ελευθερία πεπιθήσεων ε, αμφισβητείται. Έρχεται σε επαφή με τις εθνικές αρχές, θεσμικά όργανα, ΜΚΟ, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικού ηγέτες ε, και κοινότητες έρχεται σε διάλογο μαζί τους και προάγει το σεβασμό της διαφορετικότητας. Ξέρω ότι επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια, αλλά αυτό κάνει. Και είναι και ειδικό σύμβουλο προ τον Επίτροπο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία. Δεν είναι εδώ βέβαια ο Ευρωβουλευτή που έθεσε το ερώτημα, αλλά αυτή την απάντηση μπορώ να του δώσω. Θα επανεξετάσω την εντολή αυτού του ειδικού απεσταλμένου για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί. Προφανώς και το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, πρέπει κάποιος να το αναλάβει, αλλά θα το διαρευνήσω γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει ακριβώς τέτοιος ειδικός απεσταλμένος. Την επόμενη φορά μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Το άλλο σημαντικό ζήτημα που θίξατε είναι οι επιχειρήσεις και τα θέματα δικαιώματα. Σίγουρα είναι μείζον ε, ζήτημα. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, οι καταναλωτές στη Δύση με τα χαράς καταναλώνουν ε, φθηνότερα προϊόντα χωρίς να δίνουν και μεγάλη σημασία για το στο πώς ακριβώς ε, καταφέραμε να έχουμε τόσο χαμηλή τιμή. Μας νοιάζει μόνο ακριβώς να είναι κάτι φθηνό, όχι τόσο η διαδικασία. Και δεν μας ενδιαφέρει τόσο το ότι δεν ε, τηρούνται και δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους όπως απαιτούμε στην επικράτειά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα ασχολείται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη έχουμε δεσμευτικά προγράμματα σε τομείς, για παράδειγμα, εμπόριο διαμαντιών, άλλων ε, ορυκτών από ε, εμπόλεμες ζώνες, ε, αλλά και κατά των εκτελέσεων μέσω ένεσης και υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού. Και στην Ασία και στο, στις χώρες του Ειρηνικού έχουμε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα με επενδύσεις πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα προγράμματα έχουμε και στη Λατινική Αμερική. Βέβαια πρέπει να κάνουμε περισσότερα να διαμορφώσουμε την απαραίτητη συνένεση και να έχουμε την κατάλληλη εντολή για να κάνουμε περισσότερα. Έτσι βασιζόμαστε στο ε, δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Πρέπει να το αξιοποιήσετε αυτό το δικαίωμα. Και εμείς φυσικά θα σας ε, βοηθήσουμε. Έχετε όμως δυνατότητες, πρέπει να τις ε, εκμεταλλευτείτε. Γιατί όπως γνωρίζετε εγώ απλώς εκπροσωπώ ένα σώμα που μάλιστα δεν συμφωνεί πολλές φορές σε πολλά ζητήματα. Για να έχουμε λοιπόν εντολή, θα ήταν πολύ ωφέλιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να αξιοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχει, ε, προκειμένου να έχουμε μία ε, δεσμευτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως αυτό είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα ανά τον κόσμο. Άλλα ζητήματα που θίξατε. Πολλά και διάφορα. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Δέωση Επιμέλεια. Πράγματι, υπήρξε τέτοια έκκληση κατά την προηγούμενη θητεία. κρατημέλη όπως όπω η Γαλλία και οι κάτω χώρε, έχουν υιοθετήσει εθνική νομοθεσία σε αυτό το πεδίο. Άλλοι όμω όχι. Και πάλι, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα τέτοιο ζήτημα, όπου υπάρχει ισχυρή διαφωνία απόψεων μεταξύ κρατών μελών, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε.